Okay, that's quite useful. So, um, Λοιπόν, μόλις μου είπαν ότι από εδώ και πέρα οι κατάλογοι των ψηφοφοριών θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα την ίδια στιγμή που αποστέλλονται στα μέλη. Μερικές φορές γίνονται κάποιες περαιτέρω συζητήσεις γύρω από τη σωστή θέση κάποιας τροπολογίας, σαν παράδειγμα είναι κάτι το οποίο δίδει στους εμπλεκομένους κάποιες μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης και ομιλίες. Νομίζω ότι όλα αυτά πράγματι βοηθούν το να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Λοιπόν, σας καλωσορίζω, δεν θα καθυστερήσουμε άλλο. Θα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις σε εξωτερικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο των εμπορικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας. Λέει η κυρία Τσαράντσοβα. Δεν θα σας διαβάσω τη γνωμοδότηση, αλλά να μου επιτρέψετε να δώσω κάποιες εξηγήσεις. Τα PNPs, οι, οι εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού τομέα και δημόσιου τομέα είναι θέματα γνωστά. Η αρχική, ο αρχικός τίτλος της Επιτροπής ΣΥΝΚΟ ήταν κάτι το οποίο διέφευγε των αρμοδιοτήτων μας αλλά χάρη στην αστραπιαία παρέμβαση της Προέδρου μας αυτό διορθώθηκε. Τα PPPs λοιπόν χρησιμοποιούνται και στις σχέσεις της οικονομικές με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στα αναπτυξιακά προγράμματα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο εκφράζει τις επιχειρήσεις τις ευρωπαϊκές οι οποίες συμμετέχουν αρκετά συχνά στα PPPs. Οι κανόνες λοιπόν της εσωτερικής αγοράς ισχύουν η εσωτερική αγορά νομίζω είναι κάτι το οποίο τροφοδοτείται από τέτοιου είδους ε, εταιρικέ σχέσεις και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη άλλων χωρών στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τα αναπτυξιακές μας πιστώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μετέχει και αυτό θα πρέπει να γίνεται με ένα δίκαιο και ισόρροπο τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η σύντομη γνωμοδότηση καλύπτει αυτές τις λεπτομέρειες και μπορεί οι πολιτικές ομάδες να με υποστηρίξουν. Um, the shadow from the EPP is Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σκιώδης είναι ο κ. Ζωσάτη, ο οποίος δεν είναι παρόν για τους σοσιαλιστές στον Κραπίνη που δεν είναι εδώ ε, και γενικά δεν βλέπω κανέναν άλλο σκιώδη προς το παρόν για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Ναι, θα ήθελα να ε, εκφράσω ορισμένες σκέψεις της σκιώδους εισηγήτριάς μου, της κυρίας Μακλόρκιν, ο κύριος Ντόλτον. Αυτό ε, είναι μια πρόταση η οποία έγινε στην αρμόδια Επιτροπή από τον συνάδελφο της πολιτικής μου ομάδας, τον κύριο Ζαχραντήλ. Τα PPPs είναι πράγματι ένα βασικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη διεθνή οικονομική ανάπτυξη και μπορεί να βοηθήσει και την ανταγωνιστικότητα και τις καινοτομικές τεχνολογίες. Βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κερδίσουν περαιτέρω διεξόδους στις διεθνείς αγορές μέσω των κατάλληλων μορφών επένδυσης. Ε, απαιτούνται βέβαια βασικές αρχές ε, σωστής διακυβέρνησης, απαιτούνται ε, αρχές οι οποίες σέβονται τη διαφάνεια και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών στα πλαίσια της συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ε, θα προετοιμάσουμε κάποιες τροπολογίες ε, και θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας για αυτήν την ε, εισήγηση η οποία είναι πολύ σημαντική για την ομάδα, την ομάδα των συντηρητικών. Κύριε Νίλσον, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μιλήσω δανέζικα εφόσον έχω τρία λεπτά. Και εγώ πιστεύω ότι η γνωμοτοτήση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ θετικό ότι και εμείς ε, ως Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς είμαστε στην αρμόδιοι για τις συμπράξεις αυτές ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Επί της ουσίας, το θέμα είναι ο ρόλος που διαδραματίζουμε στην κοινωνική οικονομία στη Σουηδία και σε πολλές άλλες χώρες ο τομέας αυτός ε, της κοινωνικής οικονομίας είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε να τονώσουμε. Πρόκειται για ένα τομέα, για ένα τομέα ο οποίος ε, βασίζεται σε ιδρύματα, σε συνεταιρισμού και άλλες μορφές ενώσεων. Το θέμα λοιπόν είναι να προωθηθούν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις όπου υπάρχει κοινή ιδιοκτησία και καλό λοιπόν είναι να το αναφέρουμε αυτό το στοιχείο. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να απευθύνω μια παράκληση. Βλέπουμε ότι κυρίως ε, στις πιο φτωχές χώρες πολλοί κόσμος ε, φοβάται. Φοβάται όταν υπάρχει παρουσία μεγάλων επιχειρήσεων, εταιριών που αγοράζουν τα πάντα. Και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή της κοινή ιδιοκτησίας υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να γίνει μια αναφορά σύντομη και για τον κλάδο αυτό. Ευχαριστώ. Θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα δικαθιστώ τον συνάδελφο Ροζάτη, ο οποίος δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση, καθότι συνεδριάζει παράλληλα και μια άλλη επιτροπή. Αλλά και αυτός και εγώ πιστεύουμε ακράδαντα ότι το θέμα της ε, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το θέμα αυτό τίθεται στα πλαίσια της γνωμοδότησης ε, αυτής. Ο κύριος Ρωσάτη θα ήθελε να τονιστεί το εξής. Οι συνεργασίες δημοσίου και δυτικού τομέα παίζουν μεγάλο ρόλο για την ανάπτυξη και ως εξ τούτου θα πρέπει να θέσουμε τη σημασία τους για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τις εξωτερικές αγορές, τις τρίτες αγορές με τις χώρες εκείνες με τις οποίες έχει συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι συμβάσει ε, συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι μακροχρόνιες συμβάσει και θα πρέπει να διαμορφώνονται σε ένα σταθερό πλαίσιο. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες να συμβάλλουν αυτές οι συμβάσεις στην γενικότερη σταθερότητα. Επισημαίνουμε επίσης ότι το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ως το στόχαθρο την ε, ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει κοινή αντίληψη σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες που έχουν σχετική νομοθεσία, υπάρχουν όμως και κράτη τα οποία δεν έχουν διαμορφώσει νομοθεσία για τα ζητήματα αυτά και οι απόψεις επίσης διήστανται, όπως και οι στάσεις των διαφορών κυβερνήσεων και κρατών. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, θα πρέπει στο μέλλον να σκεφτούμε κυρίως την ενιαία εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά τη συμπράξη δημοσίου και δικού τομέα για την ευρωπαϊκή ελεκλήρωση. Ο κ. Ροζάτη θεωρεί ότι όταν θα ολοκληρωθεί η έκθεση θα μπορέσει να καταθέσει και αυτό στις προσωπικές του τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. So, Mrs. δεν είναι εδώ. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο για αυτή την έκθεση. Κανείς. Η Κομισιόν. Έχουμε τον κύριο Χάιερ, ε, ο οποίος είναι θεματάρχης. Ε, θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Γέσεν, τμήματάρχης από τμήμα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Αυτό είναι το σωστό όνομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τις προτάσεις ψηφίσματος. Επειδή χάνει μια ισορροπία, από τη μία αναγνωρίζει ότι οι συμπράξεις αυτές είναι μέσα για την οικονομική ανάπτυξη και από την άλλη αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν μακρά εμπειρία και γνώση σε αυτόν τον τομέα. Κυρίως Σημαντικό είναι να κάνουμε περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε ότι οι διακρίσεις που προωθούν ορισμένε χώρες αντιμετωπίζονται όταν, παραδείγματο χάρη, κάνουμε εμπορικέ συμφωνίες με αυτές τις τρίτες χώρες. Καλωσορίζουμε λοιπόν σε μεγάλο βαθμό το προτινόμενο κείμενο και περιμένουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο επί του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Θέλετε να συνοψίσετε. Δεν θα συνοψίσω, λέει η κυρία Σαράντζοβα. Συμφωνώ με τα περισσότερα από τα σχόλιά σας και περιμένω και τις γραπτές τροπολογίες σας, ούτω ώστε η γνωμοδότησή μας να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα πριν τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Everybody, we're having a Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε με διάφορους τρόπους να απλοποιήσουμε τις ψηφοφορίες μας ακόμα περισσότερο σήμερα. Έχουμε έναν μεγάλο κατάλογο ψηφοφοριών και δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο. Σενάλοβα, για το σύστημα e-call. Είναι η πρώτη έκθεση σε δεύτερη ανάγνωση που πρέπει να υιοθετήσουμε. Αρκετοί δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Συγχαρητήρια στην κυρία Σενάλοβα. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Λόπες Ιστούρις White για τις εγκαταστάσεις με σηματόσχημα, τα λοιπά. Έχουμε και τον εισηγητή εδώ, ε, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. 21. All 21. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 1.52. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 22, 23, 24 και 25 ομαδών. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 26 υπέρ. Κατά αποχή δεκτή. Πρώτη σκέψη. 1 υπέρ κατά κατά 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 154 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή ομαδών 31, 32 και 33. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απέτυχε. 156 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 34. Έχει ε, καταπέσει. 25, 26, 27 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές, 157 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 38 υπέρ κατά Α, έχει καταπέσει. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 158 υπέρ κατά αποχές δεν γίνεται δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 159 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 159. So it's 159. 159 ψηφίζεται. δεν έγινε δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 160 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 161 υπέρ κατά αποχές ε, απερίφθη. 40 υπέρ ή μάλλον 44 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή, 162 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 163 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 164 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 165 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 166 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 167 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 167. Απερίφθη. 51 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 168 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 169 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 170 υπέρ κατά αποχές απερίφθη με την ίδια πλειοψηφία 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 171 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 56 και 57 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 172 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 173 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τώρα μια μεγάλη ομάδα από το 60 μέχρι το 74. 60 με 74 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 175 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 176 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ε, ομαδών τώρα πάλι από την 76, την 77, την 78, την 177, την 178 και την 81. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. Τροπολογία 79. Α, έχει καταπέσει. 79, 80, 82, 83 και 84 έχουν αποσυρθεί. Η 179 τώρα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 180 έχει αποσυρθεί. Τώρα ψηφίζουμε 85 και 86 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 88 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 181 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 91 μέχρι και 99, 91 μέχρι και 99, υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Τροπολογία 100, με 106 συμπεριλαμβανομένης υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 107 με 115 υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 116 με 122 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 123 με 141 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Και τώρα περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 143 υπέρ για μια στιγμή. Είναι προσθήκη η 143 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 143. Λοιπόν δεκτή η 143. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 144 έχει αποσυρθεί. 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 146 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς την λέξη κατασκευή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το δεύτερο τμήμα για τη λέξη κατασκευή υπέρ κατά αποχές έχει απορριφθεί. 147 γλωσσική τροπολογία. 148 υπέρ κατά αποχές έχει καταπέσει. Η 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 6 υπέρ κατά αποχές Η, δεκτή έγινε η 5 έγινε δεκτή, συγγνώμη, η 6 λοιπόν, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 149 έχει αποσυρθεί, η 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 150 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 151 χωρίς τη λέξη ε, εργάτες της οικοδομής, εργαζόμενοι στην οικοδομή, υπέρ κατά αποχές δεκτή, ε, το δεύτερο τμήμα της 151 εργαζόμενοι στην οικοδομή υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 151. έχει απορριφθεί. Λοιπόν, τροπολογία 12 έχει καταπέσει. Τροπολογία 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20 από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Και τώρα ε, συνολική ψηφοφορία στην πρόταση ψηφίσματος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίζεται. Δεκτή. 35 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Τώρα δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε και την ψηφοφορία ε, για να δώσουμε εντολή στον Ιστούρις White για να διαπραγματευτεί εκ μέρους μας τον τριμερή διάλογο. Υπέρ, ηλεκτρονική ψηφοφορία για μια ακόμη φορά για την επίδοση εντολής στον κύριο Ιστούρις White. με την ίδια πλειοψηφία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Um, η επόμενη ψηφοφορία είναι η έκθεση για κονσάρι για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνιακών και γεωργικών ρυθμίσεων. Μεγάλος τίτλος. Και σύντομη ψηφοφορία, γιατί είναι μία και μόνη ψηφοφορία για την υιοθέτηση του αποτελέσματος του τριμερούς διαλόγου. Θα το κάνουμε, θα αποφασίσουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα. Okay. Um, Would you like to Περνάει 33 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια Λίσσα για Κονσάρη για την ψηφοφορία αυτή. Και τώρα... Ψηφίζουμε την έκθεση Κάρας για το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και αποδοτικότητας της νομοθεσίας ΡΙΦΗ, τρέχουσα κατάσταση της, ε, και προοπτικές. Είναι η, η γνωμοδότηση καρά σε αυτή την έκθεση. Συμβασμός 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, όλοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 8 υπέρ κατά αποχές. Όχι συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά. Το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Το αυτό. Καταπίπτει. 23. CP1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω καταπίπτει, αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Καταπίπτει. 26 έχει καταπέσει και πάμε στην 27 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, 28 με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε και την τροπολογία. Όχι, εγκρίνεται ούτως ή άλλως. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 40 με ναι, προφορική τροπολογία και ψήφο κατά τμήματα. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα τη 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συν όχι. Έχουμε την επιπλέον τροπολογία 42 υπέρ, κατά. Αποχές, καταπίπτη. 48 υπέρ, κατά. Αποχές, καταπίπτη. 49 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά. Αποχές, όχι. Συμβιβασμό 7 ήταν αυτό. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχέ καταπίπτει. 61 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχέ καταπίπτει. 62 υπέρ, κατά, αποχέ καταπίπτει. 63 υπέρ, κατά, αποχέ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 63. εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, το ελέγχουμε τηλεφωνικά. 64 δηλαδή νομίζω ότι εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Θέλετε να ελέγξουμε την 65 ηλεκτρονικά. Την ελέγχουμε. Έχει καταπέσει. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται ψηφίζουμε την τροποποιημένη γνωμοδότηση με ονομαστική ψηφοφορία. Οι 24 ψήφοι υπέρ, 12 αποχές, 3, 12 ε, ψήφοι κατά, συγγνώμη, 3 αποχές. Ε, περνάει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε συγητή. Και τώρα πάμε να ψηφίσουμε την έκθεση, την γνωμοδότηση Γκάλ Πέτς για την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, απολογισμούς και μελλοντικές προκλήσεις. Um, Η τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά.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 24, 24 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 26. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Ε, μάλλον δεν εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρέπτεται. 31. Υπέρ. Η 31. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Ναι, όντως εγκρίνεται. Η 53 εγκρίνεται. Η 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 55 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές καταπίπτει, ε, απορρίπτεται. Η 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά Αποχές. Έγκρινεται. 8 υπέρ. Υπέρ για την 8. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα ηλεκτρονικό έλεγχο για το 12. Εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε παρακαλώ ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Τρεις ψήφοι υπέρ, δύο κατά, τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Thank you. Um... Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τους συζητητές. Και τελευταίο θέμα στην ε, ημερήσια διαταξή για τις ψηφοφορίες. Η γνωμοδότηση της φίλης Χουσμινόβα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. και τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Όχι. Τροπολογία 1. Διορθώνει πρόεδρο. Υπέρ, κατά, αποχέ, καταπίπτει. Συμβασμό 2. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχέ, καταπίπτει. 5. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά αποχές καταπίπτει, 11 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 έχει αποσυρθεί, 14 υπέρ κατά ελέγχουμε Καταπίπτει. Συμβασμι... Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 έως 23. Έχουν αποσυρθεί όλες αυτές. Πάμε λοιπόν στην 24. Υπέρ, κατά, αποχές, Καταπίπτει. 25. 25-27 έχουν αποσυρθεί, άρα πάμε 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 29. Από... Έχει αποσυρθεί. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ κατά αποχές πίπτη 38 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 40 αποσύρεται 41 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 42 υπέρ κατά μπορούμε να την ελέγξουμε 42 έχει καταπέσει λοιπόν. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπέπτει. 48 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 48. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 54 έχει αποσυρθεί. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. 58 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές κάτι μου διαφεύγει. Μιλάω για την 64. Εγκρίνεται όμως. Συγγνώμη. Έχει περάσει. 65 και 71 έχουν αποσυρθεί. 72 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά. Παρακαλώ, 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 76 υπέρ κατά αποχές 77 αποσύρεται, 78 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. 79 με μία προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, όχι καταπίπτει, 81 υπέρ, κατά, αποχές καταπίπτει 82 υπέρ κατά αποχές νομίζω καταπίπτει να την ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά καταπίπτει όντως πολύ ωραία ψηφίζουμε το σχέδιο πνομοδότησης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Και προσθέτουμε μία ψήφο. 32 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Ευχαριστώ τη Γραμματεία και τους βοηθούς και συμβούλους που δούλεψαν πολύ έντονα για να ετοιμαστεί αυτή η λίστα, αυτός ο κατάλογος ψηφοφοριών. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Σαρανζοβά για τις συστάσεις, τις, τις τροπολογίες μάλλον, αλλά δώσουμε λίγο χρόνο για να φύγει ο κόσμος. Δίτα, θες να ξεκινήσεις λίγο. ας ξεκινήσουμε και 20, ούτως ώστε να δώσουμε χρόνο να αδειάσει η αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση της Δίτα Σαραντζόβα στις και 20. Shall we restart, um, having caught up significant amount of time? The next item on the agenda. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η γνωμοδότηση Σαρανσόβα για τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, Συμφωνία Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης εμπορίου και επενδύσεων. 266 είναι οι τροπολογίες που έχουν κρατωθεί. για την έκθεση της ε, Επιτροπής Εμπορίου, της οποίας είναι αρμόδιος ο Βέλεν Λάγκερ. Το λόγο λοιπόν έχει η συγκεκριά μα, η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω όλου του κοιόδου συζητητέ και τα, τους Συναδέλφου του υπόλοιπου που κατέθεσαν τόσε πολλέ τροπολογίες για την γνωμοδότηση αυτή. όπω είπατε, πάνω από 200 στον αριθμό ήταν οι τροπολογίε που λάβαμε από όλες τις πολιτικέ ομάδε για όλες τις παραγράφου. Προφανώ λοιπόν αυτή η συμφωνία TTIP για την εταιρική σχέση εμπορία και επενδύσεων είναι ένα θέμα φλέγων. Να τονίσω ότι το μεγαλύτερο μέρο των τροπολογιών αυτών είναι θετική ε, φύση και υπέρ τη συμφωνία. Είμαι βέβαιη λοιπόν ότι τελικά η Επιτροπή μας θα αποφανθεί ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην, ε, στις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και ότι υποστηρίζουμε τον απότερο στόχο των διαπραγματεύσεων όπως αναφέρεται στην εντολή διαπραγμάτευσης. Φυσικά υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις τώρα σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες των τροπολογιών. Εγώ με τους Κιώδης ξεκίνησα την κατάρτιση συμβαστικών τροπολογιών. Έχουμε συμφωνήσει με πολλούς επί της αρχής και ο τελικός κατάλογος θα είναι έτοιμο στο τέλη της εβδομάδας. Κάθε συμβιβασμό επιχειρεί να ισοσκελίσει τα διάφορα συμφέροντα των διαφορών ομάδων και ως εισηγήτρια έχω δεχτεί κάποια κομμάτια από μερικές τροπολογίες τις οποίες δεν θα υποστηρίζα όπως θα φανεί και από τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Ελπίζω λοιπόν τα μέλη να σεβαστούν τους συμβιβασμού όπως έχουν συμφωνηθεί στο κατάλογο ψηφοφοριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες τροπολογίες δεν θα τις ε, εξετάσουμε μία προς μία, γιατί είμαι βέβαιη ότι οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να τονίσουν ποια είναι τα βασικά μηνύματα σε κάθε τροπολογία. Θα ήθελα ανταυτού να εξηγήσω τη γενικότερη προσέγγιση που θα ακολουθήσω και στις συστάσεις. Θα ήθελα καταρχάς να καταψηφίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες που είναι εκτός της αρμοδιότητας της Επιτροπής ΙΜΚΟ ιδιαίτερα δε βουλευτών που δεν είναι μέλη της Επιτροπής αυτής. Ακόμα και αν συμφωνώ επί της αρχής και επί του περιεχομένου με κάποιες εξ αυτών, οι τροπολογίες αυτές δεν ευνοούν την ε, λήψη υπόψη της γνωμοδότης μας ε, από την Επιτροπή ΙΝΤΑ. Θα ήθελα να μείνουμε εντός του πεδίου αρμοδιότητων μας. Για παράδειγμα, όλες οι τροπολογίες για το ISDS θα σημειωθούν με αρνητικό πρόσημο. Να σας διαβεβαιώσω ότι θα γίνει μεγάλη συζήτηση στην ίντα για το θέμα αυτό και στην Ολομέλεια εκ των υστέρων. Ενδεχομένω και μια πιο σύγχρονη η ΕΣΔΕΣ. Εκ παραλλήλου ξέρω ότι ανεξάρτητα από αυτά που αναφέρονται στο κείμενο της ΕΜΚΟ, δεν θα συμπεριληφθούν αυτά στο κείμενο της ΙΝΤΑ, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου όσο και ένθερμα να το συζητήσουμε, δεν θα ληφθούν υπόψη τα σημεία αυτά από την δική μας Επιτροπή. Να το λάβουμε λοιπόν αυτό υπόψη και σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του κατάλογου ψηφοφοριών. Κατά δεύτερον, είναι προς το συμφέρον μας να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη αυτή η γνωμοδότηση για να ληφθεί υπόψη από την ίντα. Με 14 γνωμοδοτήσεις είναι πολύ πιο πιθανόν τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου να λάβουν υπόψη ένα πιο σύντομο κείμενο παρά ένα κείμενο το οποίο περιλαμβάνει γενικολογίες και επαναλήψεις. Θέλω λοιπόν ένα κύριο μήνυμα να συμπεριλαμβάνεται στην δική μας γνωμοδότηση πρωτότυπο. Και επίσης να μην υπάρχουν αντιφατικές τροπολογίες. Δεν πιστεύω για παράδειγμα ότι χρειάζεται να μπαίνουν ακριβώς οι ίδιες προτάσεις και φράσεις σε κάθε παραγράφος. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε εύστοχοι και σύντομοι στη γνωματοδοτησή μας. Μάλιστα. Άρα ε, κάπου εδώ θα σταματήσω και προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. 226 τροπολογίες δεν είναι και κανένα ρεκόρ βέβαια αλλά είναι ένα σημαντικός αριθμός. Σας ευχαριστούμε πάντως για τις εξηγήσεις σας. Αντί για τον κύριο Σφάμπ, κυρία Πέλτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Σφάμπ δυστυχώς βρίσκεται σε αποστολή και ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Θα μεταφέρω λοιπόν τις απόψεις του σε σας. Έχει ήδη δηλώσει κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης που έγινε ότι είναι ιδιαίτερος ικανοποιημένος από την πρόταση. Εξ ονόματός του μόνο θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας στην τροπολογία 160. Ο κύριος Σβάμπ Πιστεύει ότι η δημόσια ακρόαση η οποία οργανώθηκε ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και μας έδειξε ποιες είναι οι προκλήσεις. Ο κύριος Σβάμπ θέλει να συνεχίσει την συνεργασία με τον εισηγητή έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα διατύπωση και να καταστεί έτσι το κείμενο πιο αποδεκτό. Για την 120 ο κύριος Σβάμπ Ε, υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει η τροπολογία αυτή να περιορίζει τις επιλογές ε, του παροχέα. Και αυτό αφορά τις υπηρεσίες. Δεν μπορεί λοιπόν ε, να καλύπτονται οι υπηρεσίες οι οποίες επιλέγονται από μία πλευρά της σύμβασης μετά το πέρας της χρονικής ισχύως ε, του συμβολέου, της συμβάσεως. Ο κύριος Σβάμπ άλλωστε ήρθε σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίοι συμφωνούν με τη συγκεκριμένη εξαίρεση. Για τις τροπολογίες 112 και 96 επίσης, εδώ ο κύριος Σβάμπ θεωρεί ότι ό,τι έχει σχέση με τις δημόσιες προμήθειες και το θέμα των εκχωρήσεων ε, που έχει συζητηθεί τελευταία θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται ε, στο περιεχόμενο της πρότασης. Είναι πάντα στη διάθεση της εισηγήτριας ο κύριος Βάμπα ε, για μια καλύτερη διατύπωση των συμβιβαστικών τροπολογιών 4 και 6. Θεωρεί ο κύριος Σβάμπ ότι είναι αποδεκτές όλες οι υπόλοιπες συμβιβαστικές και η συγγήτρια μπορεί να ε, στηρίζεται ε, στην, στον κύριο Σβάμπ για περαιτέρω μορφές συνεργασίας. Σέλντε Μόζα στη θέση της Γκέπχαρτ. Δυστυχώς η κυρία Γκέπχαρτ δεν είναι εδώ σήμερα. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για μια εξαιρετική δουλειά και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια καλή ε, συμφωνία στα πλαίσια της ΣΥΝΚΟ. Ε, μου έχει μεταφέρει ορισμένες σημειώσεις η κυρία Γκέπχαρτ. όχι για τις συγκεκριμένες τροπολογίες αλλά για τις βασικές αρχές που θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρόταση αυτή. Καταρχάς είναι παράδοση για την σοσιαλιστική ομάδα να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε το TTIP να είναι προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών και πολιτών και εργαζομένων. Έχει μεγάλη σημασία για την ομάδα μας στον τομέα των υπηρεσιών το δικαίωμα ρύθμισης και ελευθερίας κίνησης, ελευθερίας κίνησης που έχουν οι συμβαλόμενοι να μην περιορίζεται. Ε, όμως ε, στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών πρέπει να πούμε εφόσον δεν εξαιρούνται από τις διαπραγματεύσεις πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ το συμφέρον των ε, Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την συνεργασία σε επίπεδο νομικό. Ε, πρέπει να συνεχίζουμε σε υψηλό επίπεδο κάθε προσπάθεια προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών και θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ο κανόνας της χώρας προέλευσης που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Τέλος, θεωρούμε ότι ένα TTIP αν δεν καλύψει και τον τομέα των δημοσίων προημήθειών δεν θα έχει μεγάλη ωφέλεια ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν κάποιες λύσεις στις διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Και τέλος για μια ακόμη φορά για μας, για την πολιτική μας ομάδα, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα, στα συμφέροντα τα οποία εμφανίζονται εδώ προς όφελος ε, κυρίως των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών. Τότε θα έχουμε πετύχει. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Για την κυρία Μακλάρκιν θέλει να πάρει κάποιο το λόγο. Ο κύριος Ναι, είμαι σκιώτης. Είμαι σκιώτης. Ναι, αν θέλετε να ανανεώσουμε το κατάλογο των σκιωδών. Θέλουμε καλύτερη επικοινωνία στο ιστορικό της ομάδας. Από δική μα πλευρά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, δουλειά που έχει κάνει. Για μία γνωμοδότηση, για μη νομοθετική πρόταση είναι πολλέ αυτές οι τροπολογίες και αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει τη σοβαρότητα του θέματος για την Επιτροπή μας και πόσο ευάλωτη και δέστητη είναι κάποιοι αυτού του τομεί που θα αγγίξει το TTIP. Συμφωνώ εν γέννη με τη θέση της εισηγήτριας σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που δεν εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητων της Επιτροπής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλουμε να έχουμε επιρροή στους τομείς εκείνους όπου έχουμε αρμοδιότητα, να μην αποδυναμώσουμε την γνωμοτοδησή μας με άσχετα στοιχεία σε ό,τι αφορά τον τομέα αρμοδιοτήτων μας. Να επικεντρωθούμε σε αυτά που απασχολούν εμάς, για τη θέση μας ως ομάδα. Μας ικανοποιούν οι συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύουμε ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των συμβαστικών τροπολογιών αυτών η συγγήτρια. Έχουμε ένα θέμα στην συμβαστική 10 σε ό,τι αφορά τη φράση sectors covered by the agreement, στους τομείς που περιλαμβάνονται από τη συμφωνία. Εδώ έχουμε μια μικρή αμφιβολία, αλλά εν γέννη πρέπει να πω ότι μας ικανοποιεί η κατεύθυνση που παίρνει η έκθεση, η γνωμοδότηση. Ιδιαίτερα για τους καταναλωτές, το TTIP αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία, αρκεί να προστατεύσουμε τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη. Να έχουμε μεγαλύτερη προσβασιμότητα και σε καλύτερε τιμέ σε αγαθά σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους καταναλωτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ντένις Στήλ είναι ο επόμενο. Ευχαριστώ. Παρά το γεγονό ότι ο συνάδελφο κατέθεσε πολλέ τροπολογίε. θέλω να σα πω ότι σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε τη ΕΜΚΟΥ, Δύο στοιχεία μπορούμε να θέσουμε στο επίκεντρο ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και η διαχείριση του TTIP γιατί είναι μια επενδυτική συμφωνία η TTIP αλλά ουσιαστικά δημιουργούμε μια ιστορική αγορά. Αυτή η ιστορική αγορά θα μπορούσε να διευρυνθεί και παραπέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Θα μπορούσε να συμπεριλάβει των ειρηνικών, την Ιαπωνία. Άρα θεωρώ ότι αυτή η ιστορική αγορά ουσιαστικά εξαρτάται από το TTIP. Γι' αυτό λοιπόν τα θέματα διαχείρισης του TTIP πρέπει να μας απασχολούν. Καταλαβαίνω τι λέει η συγγετρία για το ISDS ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του, της Επιτροπή μας. Αλλά το μέλλον της ιστορικής αγοράς εξαρτάται και από το σύστημα του ISDS. Το δικαστήριο, για παράδειγμα, στο Λεξεμβουργό εξέδωσε μια απόφαση το Δεκέμβριο για τη Συμφωνία Προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή στην ε, Χάρτα Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Δεν έχω δει μια γνωμοδότηση τέτοια, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα για τέτοια ζητήματα. Δεν έχουμε ε, ε, τελειωτικό κείμενο, οριστικό κείμενο για το TTIP. Μπορεί να έχουμε για το CETA, αλλά για το TTIP. Αλλά ενδεχομένω η νομολογία μας να διακυβευθεί στα πλαίσια του TTIP. Αν υπάρξει απόφαση για το ISDS που θα κινείται προ την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό έχουμε μελετήσει ποτέ αυτό. Δεν έχουμε δει ποια θα είναι η στάση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά την ε, ρυθμιστική αρμοδιότητα στο μέλλον. Η ΙΜΚΟ θα μπορεί για παράδειγμα να καταθέσει τροπολογίες σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της ε, Ρυθμιστικής ε, Επιτροπής. Κοιτώντα λοιπόν την αριθμό των συστάσεων που προέρχονται από την Επιτροπή, πέρα από το μέλλον της ουσίας της εργασίας μας, θεωρώ ότι είναι πολύ προσβεσμένο το πεδίο εφαρμογή. και γι' αυτό λοιπόν η άποψη της ομάδας μου είναι να πάρουμε στα σοβαρά το μέλλον της Επιτροπής μας, το μέλλον της εσωτερικής αγοράς. Να μην ε, αφήσουμε να μας κατευθύνουν αρχές τις οποίες δεν έχουμε εφαρμόσει ποτέ σε άλλες ε, εκθέσεις και γνωμοδίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ε, Βίκη. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια βασική διαφορά φιλοσοφική στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να αντιληφθεί την διατλαντική αγορά. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Τσαράντσοβα, για την δουλειά την οποία έκανε ε, και αυτά τα οποία μας παρουσίασε μερικές φορές ε, ξεπερνούν ή είναι και αντίθετα τις προσωπικές της αντιλήψεις. Έχει υπάρξει λοιπόν μία προσπάθεια να ληφθούν υπόψη εν μέρη τουλάχιστον οι δικές μας προτάσεις. Τώρα για το θέμα της συνεργασίας ε, και της ιδιωτικής διαιτησίας ε, σε μια επιτροπή η οποία έχει σαν στόχο την προάσπιση και της εσωτερικής αγοράς και των καταναλωτών και τον σεβασμό των κανόνων δεν μπορούμε εμείς να θεωρήσουμε ότι το θέμα της ε, διακανονιστικής συνεργασίας και της ε, ιδιωτικής διαιτησίας είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συζητήσουμε. Αυτή η διακανονιστική συνεργασία δεν μπορεί να έχει σαν στόχο να απαγορεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον να παίρνει αποφάσεις εάν δεν περάσει από την σκύλα και χάριβη της προσπάθειας κοινή θέσης με τη ΣΥΠΑ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν εναντίον της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικής μας πολιτικής. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να θεωρήσουμε ότι το θέμα αυτό είναι ένα απλό διαδικαστικό θέμα. Πρόκειται για κάτι το οποίο εντάσσεται σαφώς στις προσπάθειες τις οποίες πρέπει να κάνουμε για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και για το σεβασμό των κανόνων. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επιμείνω για μια ακόμη φορά έτσι ώστε τα θέματα αυτά να καλυφθούν πλήρως στα πλαίσια της συγκεκριμένης γνωμοδότησης της ΣΥΜΚΟ. Και έτσι και αυτά είναι θέματα τα οποία καλύπτονται και για τα οποία ενδιαφέρονται και οι ειδικοί και το κοινό. Και θα ήταν περίεργο εμείς σαν Επιτροπή να μην εκφραστούμε πάνω σε αυτά, έστω και για να προκαλέσουμε την προσοχή και να πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτού του είδους την διακανονιστική συνεργασία να περιορίζει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να νομοθετεί αυτόν αυτονόμως. Συνεπώς λοιπόν θα υπάρξει ένας μεγάλος ε, συμβιβασμός σε κάποια φάση. Ο συμβιβασμός αυτός ε, θα πρέπει να μαζέψει τα ψίχουλα που θα έχουμε αφήσει ουσιαστικά πίσω. Θα πρέπει να μας βοηθήσει να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε και ευχαριστώ τον εισηγητή που στα πλαίσια αυτής της, την εισηγήτρια που έβαλε σε αυτήν την παράγραφο την ουσία των θεμάτων τα οποία θέλουμε εμείς ε, να προωθήσουμε. Χωρίς βέβαια να καλύπτουμε το θέμα αυτό απόλυτα. Τώρα, ε, admise dans un des compromis sur la question des marchés publics, nous aimerions bien également la voir euh, sur la question des services de manière à ce que euh, nous n'ayons pas euh, de de non-retour sur un certain nombre de liberalisations. Donc, οι ε, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε σχέση και με το περιβάλλον αν θέλετε. Και εδώ τίθεται το θέμα αυτό στα πλαίσια της ε, συμβιβαστικής υπαρήθμου 3. Υπάρχουν επίσης και κάποιες μορφές οριζόντιας εξαίρεσης για τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας και της εκπαίδευσης. Πρόκειται για κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες ε, δεν είχαν έτσι και λιώς συμπεριληφθεί στην οδηγία Μπόλκενστάιν. Θέλουμε να μην συμπεριληφθούν και στη συνθήκη αυτή. Γιατί εφόσον δεν υπάρχουν στην οδηγία, πώς θα τα βάλουμε αυτά σε μια συνθήκη, γιατί θα δημιουργηθεί μια νομική ε, σύγκρουση. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο αφορά την χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ πάλι. Καλό θα είναι λοιπόν να μπορούμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τις υπηρεσίες της δημόσιας και να μην υπάρχουν εμπόδια προς την κατεύθυνση αυτή. Μακρηγόρησα. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μειώσει μόνη της τις δυνατότητες καθορισμού των κανόνων προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Ένωσης. Κύριε Τραζίνσκι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω ότι γνωμοδοτείται για τις διαπραγματεύσεις όπου σχεδόν τα πάντα αγνοούμε γιατί γίνονται και κλεισμένων των θυρών ενάντια σε οποιαδήποτε λογική διαφάνειας. Προφανώς ε, για να αφήσουμε τους συμπατριώτες μας σε απόλυτο σκοτάδι όσο περισσότερο γίνεται. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες και θεωρούμε ότι οι φόβοι μας είναι θεμητοί. Αυτά είναι υπέρ των Πολιτειών που είναι πολύ επιθετικοί εμπορικά απέναντι στι αγορές μας που δεν προστατεύονται επαρκώ λόγω της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας που κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φόβη ότι αυτή η συμφωνία ε, με νέους κανόνες ε, θα επιβληθούν σε εμά χωρί να το επιθυμούμε. Γιατί α μην είμαστε αφελεί. Πάντα ο νόμο του πιο ισχυρού επιβάλλεται στο εμπόριο. Α έχουμε την ταπεινοφροσύνη να πούμε ότι δεν είμαστε παρκώ οπλισμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων που στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι ε, αποσταθεροποιημένε από την ε, έλλειψη προστασία των δραστηριοτήτων του. Μην πιστέψετε ότι είπα ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν τι ε, προστατευτικέ πολιτικέ για τα ωραία μάτια εδώ ημών των Ευρωπαίων. Θα πρέπει να θα πρέπει να εξα... Ε, εξαιρέσουμε πάρα πολλούς τομείς. Λέτε επίσης ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν. Ε, πώς θα γίνει αυτό, ε, μόνο χάρη σε κάποιες ε, φρούτες ελπίδες, ε, για να μην ε, μας κατηγορήσουν για λαϊκισμό ορισμένοι. Ε, εγώ το λέω όλα αυτά γιατί ανησυχώ για τους ε, συμπολίτες μου, κυρίως για τους Γάλλους αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Οι περισσότεροι Γάλλοι αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι είναι κατά αυτού του, αυτού του project. Όχι γιατί είναι ηλίθιοι ή γιατί δεν το εξήγησαμε καλά, αλλά γιατί. Επειδή γνωρίζουν ε, την πραγματικότητα ε, και που, ε, την οποία πραγματικότητα εσείς πάνω στις μαλακές πολυθρόνες σας ξεκινάτε, δεν θέλουν να τη δεχτούν. Γι' αυτό λοιπόν υποβάλαμε μία τροπολογία απλή. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων και με βάση τις συνέπειες που αυτή η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα έχει στους πολίτες μας, θα ήθελα η Επιτροπή να οργανώσει ένα ρεφερέντουμ, ένα δημοψήφισμα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα, κάνετε, θα τιμήσετε εδώ το Κοινοβούλιο. Θα έχει δύο πλεονεκτήματα. Θα ενημερώσει τους συμπολίτες μας για τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, αν υιοθετηθεί. Και θα τους επιτρέψει να λύσει το πρόβλημα, να λύσει το πρόβλημα της αδιαφάνειας. Δεύτερο πλεονέκτημα θα δοθεί ο λόγος στο λαό, το αξίζει. Όχι μόνο γιατί ε, φοβόμαστε ε, ότι θα φάμε ε, μοσχάρι και βοδινό, ας πούμε, ορμόνες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί θεωρώ ότι πρέπει δημοκρατικά να σεβαστώ τις προσδοκίες όλων όσων μας εξέλεξαν. Ευχαριστώ. I'm going to start taking a speakers list. Can you signal if anybody else who would like to speak? Um, Uh, thank you, Vicky. Uh, I would like to κάνω να μιλήσει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, συγχαίρω την εισηγήτρια για την πολύ καλή τροπολογία και μου κάνει εντύπωση που έχουν τόσες πολλές. Ε, πολύ καλή γνωμοδότηση, συγγνώμη, και μου, κάνουν, μου κάνει εντύπωση που έχει τόσες πολλές τροπολογίες. Ε, επίσης, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ε, επικρίνουμε κάτι που δεν το έχουμε δει. Σε όλου του γύρου των διαπραγματεύσεων δεν έχει σημειωθεί πρόοδο. Θα πρέπει να αφήσουμε το ελεύθερο όσο μπορούμε στην Κομισιόν, ούτω ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί. Εμεί βγάζουμε όλο το φόβο μας, τον αμερικανισμό μας, το λαϊκισμό μας, τη στιγμή που το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η εντολή έχει δημοσιευτεί από την Κομισιόν οι οδηγίες από την Κομισιόν έχουν επίσης δημοσιευθεί. Ποτέ στην ιστορία εμπορικών συμφωνιών δεν έχει υπάρξει μια τέτοια δημοκρατική και διαφανής διαδικασία όπως αυτή. Και η δημόσια συζήτηση που κάνουμε σε επίσημε ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι η απόδειξη. Ε, τα σεμινάρια, οι συζητήσεις που κάνουμε, οι ακροάσεις, όπου το κοινό συμμετέχει, ακούει και κρίνει. Η δύση όμως και εξηγούμε, ε, λαμβάνουμε υπόψη μας και για την ε, ευημερία των ζώων και για την ε, διατροφική ασφάλεια κτλ. Ε, ακούμε τις, τους φόβους του κόσμου και εξηγούμε. αυτά που λέτε εσείς είναι δημαγωγική φόβη και είναι ανεύθυνο. Θέλω να συμφωνήσω με την ηθηγήτρια, θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το όραμα, την ορμή, να μην χάσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και η ανησυχία μας είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα χαλαρώσουν. Θα δώσουν ε, προτεραιότητα στη συμφωνία με την Ασία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εάν δεν συμφωνήσουμε με τον ε, μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή εμπορικό μας εταίρο που είναι η ΕΠΑ, που είναι πιο κοντά μας, με ποιον θα κάνει η συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να μιλάμε με τα χειρότερα λόγια για τα πρότυπά τους, αντί να λέμε ας πούμε ότι θα τρώμε χλώριο, ορμόνες ε, και γάματα φόμικρον, όταν ξέρουμε ότι τα πρότυπα για τα τρόφιμα δεν μπορούν να αλλάξουν με τέτοιες συμφωνίες. Μόνο από εμά μπορούν να αλλάξουν με δικά μας νομοθετήματα, όχι από εμπορικές συμφωνίες. Και η Κομισιόν για τις δημόσιες συμβάσεις, για τις δημόσιες προμήθειες, για τις δημόσιες ε, υπηρεσίες έχει απόλυτη ε, αρμοδιότητα. Γιατί λέμε ότι θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ξέρετε ότι δεν μπορεί να αλλάξει έτσι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από άλλους. Γιατί εξαπατούμε τους πολίτες μας και ξεχνάμε ότι μιλάμε για εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Αυτά είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να τους δώσουμε ε, δουλειά χωρίς να ξοδεύουμε λεφτά των φορολογουμένων, μας. Το θέμα είναι πώς θα συνομιλήσουμε με τις πολιτείες, πώς θα έχουμε θετική στάση, πώς θα είμαστε λακωνικοί ε, στο κείμενο το οποίο θα δώσουμε στην ε, ίντα και η προστασία των επενδύσεων δεν έχει τίποτα να κάνει με τις δικές μας αρμοδιότητες, είναι τεχνικό θέμα. Και στην ε, συμφωνία που έχουμε διαπραγματευτεί με τον Καναδά υπάρχουν εξαιρέσει για την υγεία, περιβάλλον και την ασφάλεια των ε, προϊόντων. Το διαβάσατε όλα αυτά. Μπορείτε να διαβάσετε, εν πάση περιπτώσει, τη συμφωνία ε, υπό τη μορφή που έχει λάθει μέχρι στιγμή. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν και υπάρχει πραγματική διαφάνεια και δημοκρατία. και ελπίζω ότι πολλέ από αυτέ τι τροπολογίε θα έχουν αρνητικό πρόσημο. Φόρντ. Θέλει κάποιος άλλος να σχολιάσει. Θέλει η Κομισιόν να σχολιάσει. Η κυρία Χουμπερ ήταν επικεφαλής, είναι επικεφαλής μάλλον τμήματος, τμήματάρχης από πλευράς Κομισιόν, δεν θέλει να σχολιάσει όμως. Ο κύριος Βανέκχαρτ από την Κομισιόν. Ο κύριος Χούμπερ. Ναι, είμαι επικεφαλής της ε, ομάδας συντονισμού πολιτικής στην Γενική Διεύθυνση Trade Εμπορίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ελπίζουμε ότι θα καταδείξουν αυτές οι τροπολογίες μια θετική ατζέντα, μια θετική στάση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που θα αφορήσει τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο κοινός στόχος όλων μας. Να σχολιάσω ένα στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε εδώ και από το οποίο θα εξαγάγουμε πολλά συμπεράσματα. Ακούσαμε την αναφορά της εσωτερικής ε, αγοράς, για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς. Αυτό αποτελεί ίσως παρανόηση του τι αποτελεί το TTIP. Είναι εμπορική συμφωνία. Έχει την κανονιστική πτυχή, προφανώς σε σχέση με τις άλλες εμπορικές συμφωνίες. Δεν πρόκειται όμως να δημιουργήσει ιστορική αγορά όπως υπάρχει η ιστορική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινού κανόνες κτλ. Κοινή νομοθεσία. Δεν πρόκειται λοιπόν να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργία ε, νομοθεσίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το TTIP. Αυτό νομίζω ότι το έχει πει κάθαρα και ένας αντιπρόεδρος. Η λήψη αποφάσεων θα παραμείνει στα χέρια των μερών της συμφωνίας. Δεν πρόκειται να υπάρξει μια μορφή διακυβέρνησης κεντρικής. Και αυτό τι σημαίνει ότι το TTIP θα διατηρήσει όλα τα στοιχεία που μας απασχολούν. Όχι μόνο το δικαίωμα νομοθεσία, οι κοινοφελεί υπηρεσίε, δεν πρόκειται να υπάρξουν δεσμεύσει σε ό,τι αφορά τι κοινοφελεί υπηρεσίε, όπω είναι η ίδρυυση, η εκπαίδευση και το θέμα της ε, ρήτρας ράτσα, της μη αναστρέψιμης ρήτρα ουσιαστικά δεν αφορά τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε όσο πιο ψηλά πρότυπα γίνεται. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούμε να υποτιμηθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. και θέλουμε και ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο εξακολουθούμε να προσπαθούμε σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την, ΣΥΠΑ και για το ISDS το οποίο αναφέρθηκε. Να υπογραμμίσω ότι η κυρία Μάλμστρομ αύριο στην Επιτροπή ΙΝΤΑ θα παρουσιάσει κάποιες προκαταρτικές σκέψεις για το πώς εμείς από πλευράς της Επιτροπής βλέπουμε την αναθεώρηση του ISDS και τέλος αναφέρθηκε ο ενδεχόμενος αντίκτυπος των αποφάσεων ISDS, των ε, επιδιδετικών ε, συμβουλίων στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το ISDS και τα επιδυτικά όργανα εφαρμόζουν μόνο τους κανόνες ε, επενδύσεων που δεν μπορούν να τους επικαλιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτό το σύστημα επιδιτησίας το οποίο εφαρμόζει μόνο τους κανόνες, επαναλαμβάνω, που ορίζονται στη συμφωνία βάσει τις οποίες έχουν ιδρυθεί και τίποτε άλλο. Θα ήθελα λοιπόν άλλη μία φορά να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την επικοδομητική σας εργασία και για το έργο που έχετε κάνει για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και εγώ θα ήθελα να μπω στον ε, κατάλογο των ομιλητών, γιατί και εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι η γνωμοδότηση έχει μείνει εστιασμένη. Γιατί αν θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά, να πάρουν υπόψη την άποψη της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να φαντήσουμε να μην είναι ευχολόγιο, αλλά να είμαστε πολύ εστιασμένοι. Αυτή είναι η Επιτροπή λοιπόν που προσπαθεί επί σειρά ετών να καταργήσει τα εμπόδια στην αγορά για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά ένθαν και ένθαν του Ατλαντικού, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως καταργώντας τα εμπορικά εμπόδια και ιδιαίτερα και τα μη εμπορικά προσκόμματα τα οποία απασχολούν πολύ τις ε, μικρές επιχειρήσεις. Το να υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι το δικό μας είναι καλά και το δικό τους κακό. Αλλά όπου μπορούμε να συγκλίνουμε για να άρουμε τα εμπόδια τα προσκόμματα στο εμπόριο, αυτό θα ήταν θετικό. Όλοι ξέρουμε ότι είναι περίπλοκη αυτή η διαδικασία και δεν πρέπει να υποτιμούμε την, ε, τις δικές μας νομοθετικές διαδικασίες και τις δικές μας κανονιστικέ διαδικασίες. Νομίζω ότι όμως πολλά μπορούμε να κάνουμε για να τονώσουμε την ε, την εμπιστοσύνη του κόσμου και επαναλαμβάνω, όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, ότι δεν πρόκειται να αντικειδεύσουμε με τη συμφωνία αυτή της κοινοφιλής υπηρεσίας την εκπαίδευση, την υγεία. Πρέπει να φροντίσουμε να τα πιστέψει η δημόσια γνώμη αυτό το παράγοντα. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και οι δημόσιε συμβάσει. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό από τη δική μα επιτροπή, γιατί οι δημόσιε συμβάσει ασφαλώ εμπίπτουν στο δικό μας πεδίο αρμοδιότητας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπίσουμε εμείς αυτό το τμήμα της συμφωνίας. Δίτα, θέλεις να σχολιάσεις και να μας πεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Κάποιοι από τους συναδέλφους έχουν ήδη φύγει. Θα έχω την ευκαιρία να εξηγήσω τις συμβαστικές τροπολογίες αυτούς στις ε, στη συνεδρίασή μας το απόγευμα. Να επαναλάβω αυτά που είπατε και εσείς και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ελπίζω αυτό το έντονο μήνυμα, το ισχυρό μήνυμα για την προστιθέμενη αξία που φέρνει η Επιτροπή μας στις διαπραγματεύσεις θα μεταφραστεί και θα απεικονιστεί και στο κείμενο. Και θα βρούμε την σωστή ισορροπία στο κείμενο. και ότι οι περισσότερες ομάδες θα μπορέσουν να συμφωνήσουν με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλους όσους πήρατε το λόγο στη σημερινή συζήτηση. Από ό,τι άκουσα, έχω την αίσθηση ότι με τις συμβαστικές τροπολογίες κινούμαστε στην σωστή κατεύθυνση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και τις ε, τελικές συμβαστικές τροπολογίες σύντομα. θα ψηφίσουμε στην έκθεση εδώ στην Επιτροπή στις 24 Μαρτίου πριν από την ψήφο στην Ίντα στις 6 και 7 Μαΐου. Ευχαριστώ. So, should we move on to the... Λοιπόν, Πάμε στο επόμενο σημείο. Στο επόμενο θέμα για κονσάρι, διαλειτουργικότητα, Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση και πολίτες. Η Επιτροπή επί είναι η Ήτρε. Εμείς είμαστε συνδεδεμένοι σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού. Κυρία Γιακονσάρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι θετική η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λύσεις διαλειτουργικές. Το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό για την ψηφιακή αγορά έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα ηλεκτρονικά εμπόδια και να μπορέσει να εξυγχρονιστεί ο δημόσιος τομέας. Στη γνωμοδότησή μου συγκεντρώνω την προσοχή μου στις βασικές μας αρμοδιότητες και σέβομαι και τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν τρεις επιτροπές εδώ, η ΙΝΤΕ, η ΛΥΜΠΕ και η ΙΜΚΟ. Εδώ είναι τα βασικά τώρα θέματα. Ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε ιδιαίτερα είναι η σχέση των πολιτών με τις επιχειρήσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει στον τίτλο, τον εξής τίτλο μάλλον, «Επιχειρήσεις και πολίτες». Προσπαθεί να δει το θέμα συνολικά και δεν περιορίζεται στη σχέση πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών. Το περιεχόμενο της πρότασης όμως δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τους τίτλους. Γι' αυτό προσέθεσα ορισμένες διευκρινήσεις νομίζω, έτσι ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να ωφεληθούν από τα μέσα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς συμπεριέλαβα κάποιες προβλέψεις που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη πρώτον τις ειδικές καταστάσεις οι οποίες ισχύουν στις μικρό επιχειρήσεις και να διευκολύνει την έβρεση λύσεων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες των πολιτών, όπως επίσης και τις κοινωνικές πλευρές της διαλειτουργικότητας. Όλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ωφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Οι εσδήποτε δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος ICE2 θα πρέπει να είναι σύμβατες με τις βασικές αρχές λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως εγγράφονται στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Η κεντρική θέση σαν παράδειγμα του χρήστη, ε, η προσβασιμότητα είναι βασικές αρχές που πρέπει να γίνουν σεβαστές η τεχνική στήριξη προς τους πολίτες από πλευράς των επιχειρήσεων θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη και η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες με παραδοσιακά μέσα και όχι μόνο αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Υπογραμμίζω επίσης την ανάγκη που υπάρχει για ε, μελλοντικές ε, επίσης ε, δυνατότητες έβρεσης λύσεων και για την λεγόμενη ηλεκτρονική ουδετερότητα. Προτείνεται επίσης μια λύση στις απορίες που υπάρχουν για τον όρο χρήστης. Ο όρος χρήστης χρησιμοποιείται σε διαφορετικά πλαίσια και πολλές φορές αυτό δημιουργεί συγχύσεις. Προσέθεσα λοιπόν ε, κάποιες διευκρινήσεις ορισμού στο άρθρο 2. Ένας χρήστης διαλειτουργικότητας σημαίνει ότι μπορεί να είναι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό, ε, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο κεντρικός χαρακτήρας σημαίνει ότι βασικός στόχος είναι ο πολίτης και οι επιχειρήσεις, ο τελικός χρήστης, end user, φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρήσεις. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η επικοινωνία και η δημιουργία γενικά συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων. Υπάρχει κάποια έλλειψη ενημέρωσης και γι' αυτό στο άρθρο 3 υποχρεώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ε, μια στρατηγική ενημέρωσης σχετικά με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο αυτό δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό απευθύνεται όπως είπαμε κυρίως στους πολίτες και στις μικρομεσαίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι εξ αρχής διαθέσιμο. Και γι' αυτό δίδουμε ένα χρονικό πλαίσιο έξι μηνών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση σε ισχύ <clears throat> αυτών των μέτρων. <clears throat> Περαιτέρω, για την εφαρμογή του ΆΙΣΑ 2, προβλέπεται διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους, ιδιαίτερος πάλι τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες ιδιαίτερα θα πρέπει να εμπλέκονται στον μέγιστο δυνατό αριθμό προγραμμάτων Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του προγράμματος ΆΙΣΑ 2 είναι κάτι το θετικό. Νομίζω όμως ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης θα πρέπει να εμπλακεί στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότηση και τι προτινόμενε τροπολογίε, λέει κυρία Παουάνοβα. Κάποιε από τι προτάσει που σα ε, υπέβαλα στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών έληφθαν υπόψη και μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλέ από τι τροπολογίε σα. Κάποια από τα βασικά σημεία τα οποία είναι σημαντικά για μένα και που εστιάζουν στις αρμοδιότητες της ΣΥΜΚΟ, όπως είπατε και εσείς, κυρία Συγγήτρια, είναι οι διατάξεις για τις ε, πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση των λύσεων που καλύπτει τις ανάγκες τους, κυρίως τη χρήση δημοσίων δεδομένων από επιχειρήσεις και πολίτες σε ό,τι αφορά την επικοινωνία ε, με τους πολίτες για τα ωφέλη των επιχειρήσεων ε, χαίρομαι που βελτιώνεται η στρατηγική επικοινωνίας με το ISA 2. Το, ο προπολογισμό του προγράμματος δεν προβλέπει μια στρατηγική επικοινωνίας, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιο έξυπνοι τρόποι για να υπερκεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, κάτι που είναι σημαντικό είναι η πρόθεση online υλικού. Είναι καλό που υπάρχει αυτό το υλικό ε, που είναι πιο εύκολο, πιο εύληπτο, σε πιο απλή γλώσσα, πιο εύκολα προσταλάσιμο ε, στα πλαίσια του προγράμματος και εμείς ως Ευρωβουλευτές μπορούμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα ε, σε συνεντεύξεις ε, ή εμπασπιτώσει μέσω των κοινωνικών media, σε συναντήσεις με τους ψηφοφόρους κτλ. Τα ωφέλη του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν ότι βλέπουμε ότι τα γραφήματα είναι πολύ χρήσιμα ε, επικοινωνιακά μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία, ειδικά αν τα χρησιμοποιούμε online, σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη που δίδεται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Ε, είναι καλές οι λύσεις. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για να ενισχύσουν την, ε, τους πολίτες, για να διευκολύνουν τους πολίτες στα ε, πρόσφατα του lifelong learning. Ε, επίσης ε, να διευκολύνουν τους ηλικιωμένους, τους άνεργους κτλ. Όλες αυτές οι ομάδες πολιτών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ισότιμα στην ψηφιακή οικονομία και να επωφελούνται από μια πιο εύκολη πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση. Κάτι που εξασφαλίζει το ΆΙΖΑ 2. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε την ψηφιακή επανάσταση. Γι' αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα ηλεκτρονικά ε, προσόντα, ε, ξεκινώντας από τη σωστή παιδεία στα σχολεία. Η τροπολογία 10, υπ' αυτή την έννοια, είναι εκτός θέματος, ε, εκτός του προγράμματος ΆΙΖΑ 2, που δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για λύσεις που καλύπτουν συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες. Σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα του δικτύου. Καλό είναι που ρυθμίζεται αυτό το θέμα, αναφέρεται αυτό το θέμα, αλλά θα έπρεπε να είσαστε πιο συγκεκριμένοι. Ποιο είναι ο ορισμό σα και τι εννοείτε όταν βάζετε μέσα αυτή την έννοια την ουδετερότητα του δικτύου. Στην τροπολογία 1 επίση. στη θέσπιση προτύπων. Μην ξεχνάμε ότι το ISA 2 δεν είναι ε, ένα πρόγραμμα για τη θέσπιση προτύπων. Το πρόγραμμα μπορεί να αμφισβητηθεί αν ακολουθήσουμε τις ίδιες διαδικασίες με τη διαδικασία τυποποίησης. Οι εξειδικεύσεις αναπτύσσονται με τις, ε, μαζί με τις κρατικές διοικήσεις και εν συνεχεία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν. Αλλά θα ήθελα η συγγήτρια να εξηγήσει λιγάκι την τροπολογία 1. Αυτά νομίζω αρκούν. Um, thank you very Ευχαριστώ οι ηγητής από τον ECR, e την, από τον ECR την ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ε, πρέπει να εστιάσουμε στην εσωτερική αγορά και στους καταναλωτές. Και η προστασία των δεδομένων είναι θέμα της LIB. Σας ευχαριστώ που υποβάλλατε τροπολογίες για τις ανάγκες ε, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάγκη συμμετοχής τους. Για να λειτουργήσει το ISA το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εστιάσει σε περιορισμένο αριθμό στοχευμένων υπηρεσιών, να αφορά τις ε, ανάγκες των χρηστών και να λαμβάνει την υπόψη η ζήτηση. Επίσης θα πρέπει ε, να υπάρχει προσθέμενη αξία στους, ε, για τους χρήστες σε διασυνοριακό επίπεδο. Όταν ήρθε ο ο Επίτροπος Άντσιπς για την ακρόασή του εδώ είχε πει οι δημόσιες υπηρεσίες καλό είναι να προσφέρονται και επιγραμμικά, online. Είναι πολύ πιο εύκολο για τους πολίτες, για τις κυβερνήσεις και είναι πολύ πιο διαφανής αυτή η διαδικασία. Συμφωνώ, αλλά για να έχουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και των καταναλωτών θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα γενικά λέει η σκιοδησηγήτρια του ECR. Επίσης, δεν πρέπει να βάλουμε τη διαλειτουργικότητα μόνο και μόνο για να έχουμε διαλειτουργικά συστήματα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ότι δεν ε, κρατάμε την ε, παλιά τεχνολογία και να λέμε να ποιο είναι το σύστημα, έτσι πρέπει να μοιάζει. Ε, γιατί είναι διαλειτουργικό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι κολλάμε στην παλιά τεχνολογία και δεν νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Και ούτε είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ποιε ιστοσελίδε, ποιε δημόσιε υπηρεσίε πρέπει να είναι διαλειτουργικέ και να δώσουμε εκεί την προτεραιότητα. Και να δώσουμε, τέλο να βάλουμε προτεραιότητε. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Παουνόβα για την ουδετερότητα του δικτύου, προσεκτικοί και εδώ πρέπει να είμαστε. Ο ορισμό που εξετάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ουδετερότητα του δικτύου εξετάζει διάφορα είδη χρηστών. Περιπίν. Ε, στο ίντερνετ έχουμε διαφορετικά είδη χρηστών. Α, ας πούμε, οι χρήστες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ευρυζωνικές. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον ορισμό της ουδετερότητας του συνδικτύου και να είμαστε σίγουροι ότι το, μέλλον, ότι το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς το μέλλον και όχι κολλάμε στην, ότι κολλάμε στην παλιά τεχνολογία. Ε, τροπολογία 41 της εισηγήτρια που λέει ότι η αξιολόγηση του προγράμματος ISA 2 θα πρέπει να έχει πληροφορίες για τα ποσοτικά και ποιοτικά ωφέλη των λύσεων διαλειτουργικότητας, ε, χρησιμοποιώντας, ε, συνδέοντας το ICT, δηλαδή την πληροφορική με τις ανάγκες των ε, χρηστών. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και την εξοικονόμηση πόρων. Ευχαριστώ. Οι επόμενοι ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητρία για την πολύ σκληρή δουλειά που έκανε στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι συμβάλλει πολύ και βελτιώνει την, προ... την πρόταση αυτή η γνωμοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ιστορική αγορά. Όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις άλλωστε λειτουργούν διαστοριακά και συχνά χρειάζεται να έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου με τις δημόσιες υπηρεσίες. Η Εστονία είναι ένα καλό παράδειγμα. Δυστυχώς οι ηλεκτρονικές διαδικασίες σε άλλα κρατημέλη εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ περίπλοκες και αυτό δημιουργεί εμπόδια. Και αυτό εμποδίζει την ε, καλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Τονίζω λοιπόν την ανάγκη να βρεθούν στο μέλλον σωστές λύσεις. Επίσης, τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Όταν χρησιμοποιούνται λύσεις διαλειτουργικότητας. Επίσης, υποστηρίζω την τροπολογία για τη στρατηγική επικοινωνία που σκοπό έχει να ενημερώσει σε ό,τι αφορά τα ωφέλη του συστήματος και τις ανησυχίες που προκύπτουν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, ιδιαίτερη κατάσταση που αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν έχουμε σκιώδη από την πλευρά της Google από τους πράσινους. Ούτε από το EFTD έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Θα ήθελε κανείς άλλος να μιλήσει. Όχι. Παρακαλώ. Η κυρία Κάλλας. Σας ευχαριστώ. Κάποια επιπρόσθετα σχόλια γιατί δούλεψα στο πρόγραμμα ΆΙΣΑ και στα, στην Επιτροπή Διαμηχανίας. Καλώς ορίζω λοιπόν ε, τα όσα μας είπε ο εισηγητή για θέματα ενημέρωση και πληροφόρηση από πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα κράτη-μέλη θεωρώ ότι θα πρέπει να δεσμευτούν για την γοργή ανάπτυξη του συστήματος στην Ευρώπη. Να ενταρρυνθεί η χρήση υπηρεσιών online. Στην Ήτρε, οι τροπολογίε μου κινούνται προς την κατεύθυνση της σημασίας καταχώρησης των απαραίτητων δεδομένων και της ψηφιακής ε, αυτής συνεργασίας. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί τον πυλώνα του προγράμματος. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες που υποβάλλουν μία φορά μόνο αυτές τις... Ε, που θα έπρεπε με το σύστημα αυτό να υποβάλλουν μόνο μία φορά τα στοιχεία. Και έτσι θα περιοριστεί ο φόρτος εργασίας και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Ίσως θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή, εφαρμογής και για τις μεγάλες κλίμακας ε, συστήματα πληροφορικής. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτό το σύστημα, το ΛΑΙΖΑ ευρεία κλίμακα πληροφορικά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή σε κάθε περίπτωση για τη δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο. Αν όχι, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν επιθυμεί να μιλήσει. Μαργκάριτα Αμπεκάση, που είναι η υπεύθυνη για το πρόγραμμα ΆΙΣΑ. Ευχαριστώ, πρόεδρε να θίξω κάποια από τα σημεία που ακούσαμε από τους αξιότιμους βουλευτές. Το πρώτο. Προφανώς υποστηρίζουμε την ανάγκη επικοινωνίας και πληροφόρησης. Αλλά ο προπολογισμό δεν επιτρέπει να ξεκινήσουμε μεγάλες εκστρατείες πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Παρόλα όλα αυτά, έχουμε οραματιστεί την ανάπτυξη εργαλείων τα οποία θα μπορέσουν να ξαναχρησιμοποιήσουν και οι δημόσιες διοικήσεις στη συνέχεια στις επαφές τους με τους πολίτες. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να είναι γενικής φύσεως, ε, αλλά και πιο ειδικά σε ό,τι αφορά ειδικέ δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης σε ό,τι αφορά την επαφή με το κοινό και τις επιχειρήσεις, τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερω. Ύστερα, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα ωφέλη και η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολλαπλά για την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας. Το πρώτο είναι ασφαλώς ότι το πρόγραμμα γίνεται μέσω δημοσίων συμβάσεων. Άρα κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση. Κατά το δεύτερον, οι συγκεκριμένοι τομή ανάπτυξης διαλειτουργικότητας Να αναφέρω για παράδειγμα τα σχετικά μετρώα, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ψηφιακή ανάπτυξη. Αυτό γίνεται και μέσω κοινοτήτων σχετικών πρακτικών που είναι ανοιχτέ σε όλους. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Ίσως λοιπόν καλό θα ήταν να τονίσουμε πιο πολύ τη συμμετοχή σε αυτές τις κοινότητες πρακτικών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από τους ακαδημαϊκούς κύκλους ο τρίτος τρόπος ε, συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προβλέπεται και ήδη έχει εφαρμοστεί στο πρόγραμμα ISA είναι οι δημόσιες ε, διαβουλεύσεις όπως και με στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας υπήρξαν κάποιες προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν. αναπτύχθηκαν. Αυτές οι προδιαγραφές, αυτά τα πλαίσια προκύπτουν από δημόσια διαβούλευση. Άρα, ο καθένας μπορεί να συμβάλλει και η συμμετοχή του να ληφθεί υπόψη για την ε, βελτίωση των πρωτογραφών και των πλαισίων. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω. Για τις παρεμβάσεις που ακούσαμε ως τώρα για το μέλλον. Ένα από τα κριτήρια και ένας από τους όρους άλλωστε για τις μελλοντικέ λύσεις είναι να αγγιηθούμε την διαλειτουργικότητα. Και αυτό γιατί αυτό θα επιτρέψει να αναπτυχθούν εφαρμογές ανεξάρτητα από τις διάφορες ε, κυβερνήσεις. Αν υπάρχει διαλειτουργικότητα μπορούμε να αγγιηθούμε ότι κάθε ε, κυβέρνηση μπορεί να αναπτυχθεί και να αναπτύξει ό,τι θέλει χωρίς να περιορίζεται στις παραδοσιακές τεχνολογίες και χωρίς να υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το στοιχείο. το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί στην ε, εφαρμογή του συστήματος. Να αποφεύγονται δηλαδή οι περιορισμοί, οι μελλοντικοί περιορισμοί μέσω τη διαλειτουργικότητα. Αυτά λοιπόν από δική μα πλευρά επί του παρόντο. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, κυρία Γιάκονσάρη, θέλετε ξανά το λόγο, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, λέει η κυρία Γιάκονσάρη. Σα ευχαριστώ για μια καλή πρόταση, επικοδομητική πρόταση. Για την τροπολογία 1 πρέπει λίγο να τη διευκρινίσουμε νομίζω. Θα δούμε τι ανάγκες θα υπάρξουν στο μέλλον και ανάλογα θα βοηθήσουμε. Πρέπει να είμαστε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται. Γιατί η τεχνολογία στον τομέα αυτό αναπτύσσεται με πολύ υψηλή ταχύτητα. Και αυτού του είδους η ευελιξία νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάποιο χρόνο για να τα επανεξετάσουμε όλα αυτά σε με την απαιτούμενη άνεση. Ευχαριστώ λοιπόν. 31 Μαρτίου. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε σε αυτά και θα τα επανεξετάσουμε στις 6 και 7 Μαΐου. Έχω μια δουλειά στις 7 Μαΐου λέει η κυρία Φόρντ, οπότε θα προεδρεύσετε λέει στην κυρία Κορατσαμπίλτ. Λοιπόν, και η κυρία Στάιλερ επίσης 7 Μαΐου και αυτή προφανώς έχει δουλειά. Σας ευχαριστώ. Uh, Τελευταίο θέμα. Διαρωτώ με βέβαια αν από το σοσιαλιστές ο Σκιώδης είναι εδώ, είναι εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που παραμένετε. Έχουμε επίσης μια αντιπροσωπεία αυστριακών βουλευτών από το Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, είναι λίγο μυστήρια αυτή η εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανονικά έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για τις επιτροπές, αλλά την εβδομάδα αυτή έχουμε μόνο δύο μέρες συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών και έχουμε επίσης και ένα τμήμα αυτό που ονομάζουμε πράσινη εβδομάδα έτσι ώστε οι βουλευτές να πάνε σε αποστολές στην πατρίδα τους. Και γι' αυτό ακριβώς πάρα πολλοί από βουλευτές αντικαθιστούν ο ένας τον άλλο και θα δείτε βουλευτές να συνεργάζονται λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας καλωσορίζω λοιπόν τους εκπροσώπους της Αυστριακής Βουλής. Το επόμενο λοιπόν θέμα είναι η ε, γνωμοδότηση για τις επιπτώσεις των εξελίξεων στις αμυντικές αγορές σχετικές με τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης. Γκάλπετς, ο εισηγητής στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η κυρία Γκόμες η συγγητρία. Εμείς εμπλεκόμεθα σύμφωνα με το άρθρο 54 και θα υπενθυμίσω στους συναδέλφους και θα με διορθώσει η γραμματή εδώ ότι στο παρελθόν η επιτροπή μας ήταν ηγέτης σε σχέση με θέματα που είχαν σχέση με τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα επαναξεταστεί τους επόμενους μήνες. Έχει σημασία λοιπόν να ενθυμούμεθα ότι μιλάμε για τις δικές μας αρμοδιότητες. Ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και δεν αμφισβητήθηκαν οι αρμοδιότητές μας όπως είπα σύμφωνα με το άρθρο 54 και σε σχέση με νομοθετικές εκθέσεις. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκάλπες λοιπόν. Ε, πρόεδρε. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε το τεχνικό πλαίσιο αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Όπως είπατε, είναι μια διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής. Δεν είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Θα διαπραγματευτώ το θέμα με την κυρία Άννα γιατί εδώ εμπλέκονται και αρμοδιότητες άλλων επιτροπών. Η επιτροπή μας αφορά, ε, ασχολείται με θέματα κατακαιρματισμού της ε, αγοράς, με αμυντικούς εξοπλισμούς κτλ. Είναι μια, ένα σχέδιο έκθεσης ιδίας πρωτοβουλία, το οποίο θα σας παρουσιάσω. Βασίζεται στην οδηγία του 2009, κάθετος 43. Ε, η οποία έχει ενσωματωθεί πλήρως στις εθνικές νομοθεσίες. Υπάρχει το, το κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά αμυντικού υλικού εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που οι κανόνες εσωτερικής αγοράς μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτόν τον τομέα για τον καλό και δίκαιο ανταγωνισμό και για να τον αυξήσουν βεβαίω τον δίκαιο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο τομέα αυτό είναι πολύ ειδικό τομέα, πολύ εξειδικευμένο. Κατά για πολλά χρόνια υπήρχε ένας κατακαιρματισμός, γιατί ήταν εθνική αρμοδιότητα. Η Κομισιόν έχει εκδώσει διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας και για να δοθεί συνέχεια στους στόχους αυτής. Σε φάση περικοπών του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ε, ζήτηση ε, και μάλιστα με σωρευτικό τρόπο. Αυτή είναι μια αποτελεσματικότατη μέθοδος για να προχωρήσουμε. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τις, ε, τους κυβερνητικούς φορείς και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τις προμήθειες, αμυντικές προμήθειες και που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να έχουν κοινά προγράμματα προμηθειών. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις και επομένως να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας, ούτω ώστε να δρέψουν και το ωφέλη της συνεργασίας με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Μιλάμε για ειδικά προγράμματα συνεργασίας, τα οποία θα προωθήσουν την αποτελεσματικότητα. Άλλες δικαιολογημένες αποκλήσεις είναι οι διμερείς προμήθειες ή προμήθειες που διέπονται από διεθνείς υποχρεώσεις. Είναι θεμητές αυτές οι παρεκκλήσεις. Γιατί η εφαρμογή της οδηγίας θα μπορούσε να θέσει ένα αμφιβόλο την ισοτιμία στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι εξαιρέσεις ε, ερμηνεύονται εν τη στενή ενία τους, τι θα πρέπει να γίνουν καταχρήσεις για να παρακαμφθούν οι διατάξεις της οδηγίας σε καμία περίπτωση. Για να μπορέσουμε επίσης να προωθήσουμε περισσότερο την εσωτερική αγορά για το αμυντικό υλικό και για να έχουμε ε, ισότιμη μεταχείριση όλων των προμηθευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μακροπρόθε, τις μακροπρόθεσμες ε, διακριτικές ε, στάσεις και τις τρευλώσεις αγοράς. Συχνά υπάρχουν ε, διατάξεις διακριτικές που υποσκάπτουν την οδηγία και που δεν εξυπηρετούν την εσωτερική αγορά. Επίσης το Συμβούλιο θα πρέπει να βάλει αυτό το θέμα στη μερίσια διάταξη και μάλιστα το συζητήσει ε, στη Σύνοδο Κορυφή. Και αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να Έχουμε τις καινοτομίες του πακέτου και να το εφαρμόσουμε και στην, ε, στο, στους αμυντικούς εξοπλισμούς, ε, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τον ειδικό του χαρακτήρα. Οι κανόνες κατά των, αδιαφανών πρακτικών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και τα μέτρα ελέγχου για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται για να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση οι δημόσιες προμήθειες και οι δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να γίνονται πιο αποτελεσματικά. Ο βασικός στόχος θα πρέπει να έχουμε ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο για τον κλάδο του αμυντικού εξοπλισμού που θα πρέπει να υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να υπάρχει και μια βιομηχανική πολιτική σχετική με τον κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω αυτή η στόχοι να ενσωματωθούν στο σχέδιο της γνωμοδότησής μου, να περάσουν και περιμένω και τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών, τις απόψεις γενικά των συναδέλφων μου και τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ. Um, so, Olga Shanlova is standing in for Sergio Gutierrez Pietro. Yes, indeed. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ο σκιώδης εισηγητής μας δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Έχουμε κάποιες, έχουμε να κάνουμε. Θα σας διαβάσω εξ ονόματος τους. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει προκαλέσει μεγάλη μείωση του αμυντικού προϋπολογισμού στις πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει επιτρέψει στο επενδυτικό σχέδιο να αποδώσει καρπούς. Πρέπει να συντονιστούν λοιπόν ε, οι εθνικοί προπολογισμοί για την άμυνα και την... Ε, για να αποφευκθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά. Να καλέσουν τα κρατη να χρησιμοποιήσουν ε, την... τα εργαλεία που προβλέπει η οδηγία 2009-81 και 43 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την αλυσίδα παραγωγής. Θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να την κατανοήσουν καλύτερα για να έχουν πρόσβαση στις ε, σχετικές συμβάσεις για την ε, άμυνα και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση στην πληροφόρηση γιατί μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά στον τομέα αυτό είναι πολύ σημαντική για την ανταγωνιστική και αποδοτική λειτουργία και για την πρόβλεψη των ε, όσων προβλέπονται στην κοινή πολιτική για την άμυνα. Η βιομηχανία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα, πολλές, ε, πολύ λίγες νέες συμβάσεις στον Ευρωπαϊκό Στρατό και η επένδυση και η ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ standing in for... Μάλιστα. Ο κύριο Ντάντον τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόφανώ. το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη γενικά δεν δαπανούν ε, επαρκή κονδύλια ή στην άμυνα. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τι ικανότητες ε, τις αμυντικές, αλλά ούτε και για την ε, βιομηχανία την σχετική. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε τι ανάγκε της μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τομέα αυτό, όπως το έκανε η συγγήτρια. Έχω κάποιε πιο συγκεκριμένε ανησυχίε, αλλά και μια γενική ανησυχία. Στην παράγραφο 5, ιδιαίτερως η ομάδα μα δεν υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση των αντισταθμίσεων, των offset. Είναι κάποια κρατημέλη που είναι πολύ ευαίσθητα. Στην παράγραφο 8, καλώ ορίζεται, ο δικό χάρτη του 2014 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα, αν χρειαστεί και εδώ ανησυχούμε. Καταρχάς, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, πρόσθετα μέτρα. Και κατά δεύτερον, πρόκειται για μια εθνική αρμόδιότητα που με φαίνει στο επόμενο σημείο, στην παράγραφο 10, όπου υπάρχει ζήτηση να δημοσιευτεί η πράσινη βίβλος για τον έλεγχο των προσιακών στοιχείων. Δεν το υποστηρίζουμε από πλευρά του ECR αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ ανησυχούμε ότι θα προσπαθήσει να ελέγξει περαιτέρω τις ε, στρατιωτικές ικανότητες των κρατών μελών. Στον οδικό χάρτη αναφέρεται η προσέγγιση, ενδεχομένως να χρειαστεί η ευρωπαϊκή προσέγγιση και ενδεχομένως να ε, πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή αυτονομία στην ε, άμυνα και την ασφάλεια και με, σε συνδυασμό με αυτά που είπε ο κ. Γιούνκερ αυτή την εβδομάδα για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, καταλαβαίνετε πόσο ανησυχούμε. Είμαστε κατά την ομάδα μα του Ευρωπαϊκού Στρατού. Θέλουμε να είναι εθνικό ζήτημα αυτό και θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταία δρανίδα κατά τη ιδέα ενό Ευρωπαϊκού Στρατού. Άρα, οποιαδήποτε απόπειρα να μπει αυτό από την πίσω πόρτα μέσω των δημόσιων συμβάσεων σε θέματα ασφάλεια και άμυνα θα μα βρει εντελώς αντίθετους. Μετά από όλα αυτά όμως να διευκρινίσω ότι ο σκιώδης μας προσβλέπει τη συνεργασία μαζί σας με επικοδομητικό τρόπο, στο βαθμό του δυνατού. Yes, here I am again. <laughs> Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Ο γενικός τόνος είναι καλός. νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για αυτό το θέμα. Γενικά συμφωνώ με την ησυχήτρια ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά στον τομέα της άμυνας, ούτως ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, βιώσιμοι και να είναι πολύ αποτελεσματική η ευρωπαϊκή άμυνα. Α, μην ξεχνάμε όμως ότι οι προμήθειες στον αμυντικό τομέα έχει πολλές ιδιαιτερότητες που συνδέονται με την εθνική άμυνα και την και όλο το πλαίσιο της ασφάλειας κάθε χώρας. Ο δικός χάρτης του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα μιλάει και επαναλαμβάνει όλα τα στοιχεία των προηγούμενων δικών χαρτών για την ασφάλεια και την άμυνα. Ε, υπάρχει θέληση για μια ενιαία αγορά αμυντικών εξοπλισμών, γιατί θα υπάρξουν και εξοικονομήσεις. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ είναι υπέρ της δημιουργίας μιας τέτοιας ε, ενιαίας αγοράς, αλλά πρέπει να σεβαστούμε την εθνική κυριαρχία και την ε, αμυντική πολιτική των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει απόλυτη ανεξαρτησία, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ενοπλές δυνάμεις του. Ειδικά μιλάω για την παράγραφο 11 της εισηγήτριας. Είπα ότι η εφαρμογή του δικαίου που έχουμε είναι πολύ πιο σημαντική από το να δημιουργούμε νέα νομοθετήματα. Όμω, φαντάζομαι ότι οι διάφορε προτάσει για την αθεώρηση τη ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να προωθηθούν για να λάβουμε υπόψη μα καλύτερα τι ευαισθησίε του τομέα τη άμυνας από τη μία και να δημιουργήσουμε πραγματική ισοτιμία από την άλλη. Θα προτιμούσα η εκτελεστική έκθεση να είχε ετοιμαστεί νωρίτερα. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις όποιες ε, εντοπισμένες ελλείψεις. Σε ό,τι αφορά τις αντισταθμίσεις. Είμαι κατά της άποψης της ηγήτριας. Το, είναι παράδειγμα, το παράδειγμα της ε, Τσεχίας δείχνει ότι μπορεί η αμυντική βιομηχανία να βοηθήσει και να αναπτυχθούν κάποιες προβληματικές περιοχές. Ε, η ακύρωσή τους θα μειώσουν την, ε, βιομηχανική, το βιομηχανικό δυναμικό κάποιων κρατών μελών. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να το αντικαταστήσει αυτό το στοιχείο, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της εισηγήτριας ότι αφορά την προώθηση της υπεργολαβίας και την υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συμπεριλαμβανομένης και της καλύτερης πρόσβασής τους στην αμυντική αγορά. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά την εισηγήτρια για την έκθεσή της. 20 όλτες από τους πράσινους και ο δισηγητής. Δεν είναι εδώ. Να εκφράσω και εγώ κάποιες γενικές σκέψεις σχετικά με το πώς εμείς μπορούμε να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά. Να βοηθήσουμε επίσης ε, και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα των προμηθειών αμυντικού υλικού και να ελέγξουμε και με διαφορετικό τρόπο το θέμα των εξαγωγών πολεμικού υλικού. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν αρκετές ευαισθησίες. Θέματα εθνικής άμυνας, σημείο 4 σαν παράδειγμα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην θέτουμε τεχνητά όρια. Θα συμφωνήσω επίσης με αυτά τα οποία είπε και η κυρία Σενάλοβα που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνοδεύει τις εφαρμοστικές διατάξεις με νομοθετικές προτάσεις. Εφόσον είναι κάτι το αποδεκτό, γιατί να μην υπάρχει μια νομοθετική πρόταση που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε την γραφειοκρατία και έχω την αίσθηση ότι ακόμα και σε αυτού του τύπου της νομοθετικές ρυθμίσεις θα μειώσουμε τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Και δέχομαι τις προτάσεις των φιλελευθέρων ότι θα πρέπει να δούμε τι λέει η έκθεση εφαρμογής πριν να πάρουμε μια τελική απόφαση σε σχέση με τον προσανατολισμό που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι παρούσα στην ε, φάση αυτή. Επαναλαμβάνω αυτά τα οποία από πριν. Για να ε, διατηρήσουμε τις αρμοδιότητές μας θα πρέπει να δείξουμε κάποια ευαισθησία στην Επιτροπή Άμυνας, γιατί τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα όπως είπαμε. και γι' αυτό υπάρχουν εξαιρέσεις πάρα πολλές για θέματα εθνικού τύπου. Κυρία Πέλτς, έχετε το λόγο πάλι. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Όπως είπα και εξ αρχής, η αρμοδιότητά μας για το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Πρόκειται λοιπόν περιορισμένο και λεπτό. Λεπτή ισορροπία που θα πρέπει να πετύχουμε. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίε που έχουμε από πλευράς εσωτερικής αγοράς. Και συμφωνώ με τους κοιόδους συζητητές ότι ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ ευαίσθητος αν θέλετε. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε εισηγητής ε, και σκιώδης εισηγητής ε, θα ήταν πιο πολύ υπέρ της σημασίας της εθνικής αρμοδιότητας. Υποστηρίζω τις ιδέες αυτές. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι παραβιάζω τα όρια αυτά. Ευχαριστώ τους κοιότητες των σοσιαλιστών για την ιδέα τους. για την προτεραιότητα στην έρευνα και την ε, συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμπεριλαμβάνεται αυτό στο σχέδιο γνωμοδότησης σε ό,τι αφορά τώρα την πλήρη κατάργηση των εξαιρέσεων. Καταλαβαίνω ενδεχομένως την ανάγκη να αλλάξει λίγο το σημείο και διατύπωση του σε ό,τι αφορά την ε, διατύπωση της πρώτης ε, φράσης. Στην πράσινη βίβλο τώρα, στο σημείο 10, αναφέρω ότι ενδεχομένω να έχει οριμάσει η κατάσταση και η συγκυρία για να υπάρξει μια πράσινη βίβλος. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει πάντα με το σεβασμό των εθνικών κυριαρχιών. Να αξιοποιήσουμε όμως την ευκαιρία αυτή που έχουμε για θέματα εφαρμογής, για την έκθεση εφαρμογής και τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Πρόκειται μόνο για μία ένδειξη για το μέλλον. Αν υπάρχουν ε, εκθέσεις ε, πρωτοβουλίας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ποιες είναι οι μελλοντικές ε, φάσεις, οι μελλοντικές ενεχόμενες φάσεις. Αυτό ήθελα μόνο να τονίσω. Σας ευχαριστώ. Αύριο θα γίνει συνάντηση των σκιωδών όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση συμβαστικών λύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Πρόεδρος, μάλιστα. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 31η Μαρτίου και η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 20 Απριλίου για την ε, έγκριση στην Επιτροπή 24 Απριλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, και έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, μάλλον η πρωινή συνεδρίαση. Θα τα πούμε στις 3 ε, το απόγευμα, όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις με την ε, κυρία Γιούροβα, την Επίτροπο, μεταξύ άλλων για θέματα καταναλωτών.